Συγκεντρωθείτε, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση να λάβουμε. Πρέπει να συνέλθει σε σώμα το Προεδρείο της Επιτροπής, ε, να εκλεγεί πρόεδρος. Η πρόεδρος μας, όπως ξέρετε, η κυρία Βαλεάν, ορίστηκε επίτροπος. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. και να εκλέξουμε νέα πρόεδρο. Λοιπόν, ίσως και ένα αναπληρωτές ο κύριος Μπλάγκα αντικαθιστά τον κύριο Κουμπίριους, ο κύριος Σαλίνη την κυρία Νίμπλερ, η κυρία Τότ τον κύριο Γκύρκ, αυτά όλα από το ΕΛΚΑ, από τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Σούτλ αντικαθιστά τον κύριο Καλέντα, ο κύριος Τσίς τον κύριο Χάιζερ, Τσορινιού, η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα αντικαθιστά την κυρία Μπέρ, Ε, κύριο Σάνσιπ, τον κύριο Φλέγκο και από τους πράσινους η κυρία Πάολος αντικαστά τον κύριο Μπλος κύριος Καρίμ ε, αντικαθιστά τον κύριο Πέξα από το ID η κυρία Μπίλκ αντικαθιστά τον κύριο Μαριανή στο ο κύριος Ρόκερ και του τον κύριο Τοσενόφσκι και στην ΚΟΕ ο κύριος Μποτέγκα αντικαθίσταται από την Κορνέλια Έρνστ. Αυτά. Έχουμε λοιπόν απαρτία. Ζητάω λοιπόν ε, τώρα υποψηφιότητες. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ από το ΕΛΚ προτείνουμε τον κύριο Μπουζόη για πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Ζωέλ Μελών θα να προτείνω ως ε, υποψήφια πρόεδρο. Σελ Μιλάν. Ζωέλ Μελάν. Συμφωνείτε με την υποψηφιότητα. Ναι. Um, Πρέπει λοιπόν τώρα να γίνει η μυστική ψηφοφορία. Έχουμε δύο υποψήφιες. Όπως ξέρετε, κάθε βουλευτής έχει μία ψήφο. Κανονικά έχουμε ΕΛΚ 18, σοσιαλιστές 15, ΡΙΝΙΟ 10, ECR 6, ΓΚΟΕ 4 και πηγή γραμμή 4 ε, και στον πρώτο γύρο. Η υποψήφια θα πρέπει να έχει απόλυτη πλειοψηφία ε, και εννοούμε ψήφους υπέρ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. μόλις ε, θυμήθηκα ότι την κυρία Μελέν θα έχουμε κόκκινο ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Μπουσόη όχι το κόκκινο κουμπί και για την κυρία Μελέν το πράσινο. Λοιπόν, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Να δούμε αν δουλεύει το μηχάνημα. Κόκκινο για την κυρία Μελέμ, πράσινο για τον κύριο Μπουζόη, λοιπόν. Το Ορίστε. Ε, αλλάξτε θέση. Ε, τα μηχανήματα όλων των υπολείπων δουλεύουν. Είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίστε, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας, όχι. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία. Ψήφισαν όλοι. Εντάξει, πέρας. Μπουσόη λοιπόν. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Πού είναι αυτό το παιδί? Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. Να κάνω μια σύντομη δήλωση. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Σας ευχαριστώ για την ε, ψήφου σας και την εμπιστοσύνη σας και σας διαβεβαιώ ότι θα εκτελέσω τα καθήκοντα του Πρόεδρου με αίσθημα ευθύνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του ΕΛΚ, τον συντονιστή τον κύριο Έλερ, την κυρία Καρβάγιο και τους ε, συναδέλφους μου από την ρουμανική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, ε, Μπόγκταν και Μπλάγκα που μας στήριξαν. Η ίδια η Επιτροπή ΙΤΡΕ είναι κατά την απόψη μου η πιο σημαντική επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Υπεύθυνη για την βιομηχανική πολιτική, την ε, πολιτική έρευνας, καινοτομίας, διαστημική πολιτική και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο η Επιτροπή μας στις ζωές των πολιτών μας. Επιπλέον, με την, ε, νέο, την νέα επιτροπή η οποία ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει η επιτροπή μας ε, να είναι στην πρώτη γραμμή στο, στην αλλαγή υποδείγματος και για να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις που έχουμε με δεδομένη την κλιματική αλλαγή αλλά και την ανταγωνιστικότητα και τις δουλειές των πολιτών. Χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική, μια μετάβαση των συστημάτων ενέργειας για να επιτύχουμε τον στόχο απομάκρυνση από τον άνθρακα, αλλά είναι επίσης σημαντικό όχι μόνο να εμπνεύσουμε τον κόσμο, αλλά να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και μια δίκαιη μετάβαση. Οπότε, να αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεργαστούμε και ως πρόεδρος θα προσπαθήσω να προστατεύσω τις αρμοδιότητες επιτροπής μας και να διασφαλίσω μια ισορροπία και ρεαλισμό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you once again. We'll take... Ε, ευχαριστώ και πάλι. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και τα ξαναλέμε στις 10.